και την τελευταία στιγμή να έρθουμε σε επαφή και να κουβεντιάσουμε πώ μπορούμε να έχουμε κοινό κείμενο εδώ στο Κοινοβούλιο για το θέμα αυτό. Ο Πρόεδρο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μήπω κάποιο θέλει να παρέμβει κατά του αιτήματο. Όχι, ούδη. Επομένω, ποιοι είναι υπέρ του αιτήματο ψηφίζουμε. Υπέρ. Ε, ευχαριστώ. Κατά. Αποχέ. Συνάδελφε. Εγκρίνεται το αίτημα και θα συζητηθεί στο τέλος των εργασιών της Τετάρτης όπου τέλος τέλος έχουμε χρόνο. Αυτά. Επομένως τακτοποιήθηκε και αυτό. Και προχωρούμε τώρα στο πρώτο θέμα το οποίο είναι η Συμφωνία Διεθνικής Σύμπραξης Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μαρόκου που είναι το πρώτο θέμα της μεσής διατάξεως. Μην φεύγετε καθίστε, μην μας εγκαταλείπετε. If you want to leave us... Εάν θέλετε να φύγετε συνάδελφοι, δεν είναι αυτό τόσο ωραίο, αλλά να το κάνετε, να το κάνετε γρήγορα. Μια ώρα αρχίτερα, προτιμούμε να κάτσετε μαζί μας and not to discuss in the hall. Όχι κουβεντούλες στους διαδρόμους. Mm. Uh, Ωραία, αγαπητοί φίλοι, αρχίζουμε τη συζήτηση. Καρλ Χάγλοντ, συνάδελφε. Είστε εισηγητή, αλλά ταυτόχρονα είστε και συντάκτη της εκθέσεως. Θέλετε να αθροίσετε το χρόνο αυτών των δύο ιδιωτήτων. Άρα, σύνολο ένα εξάλεπτο. Ναι, ναι, έχετε το λόγο. Εισηγητά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα υποφεληθώ της ευκαιρία και θα συζητήσω όπως προτείνατε και τα δύο σημεία μαζί. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω το ψήφισμα το οποίο συντάξαμε με τη συνάδελφο Κάρμεν Φράγκα. Είναι ένα ψήφισμα σχετικά με το πρωτόκολλο ελευθερικής συμφωνία με το Μαρόκο, κάτι το οποίο έχουμε συζητήσει αρκετές φορές στο Κοινοβούλιο την τελευταία χρονιά. Φτάσαμε σε μια χρονική στιγμή όπου μπορούμε να συμφωνήσουμε πολλέ ομάδε συμφώνησαν σχετικά με το περιεχόμενο του ψηφίσματο. Ξέρω ότι υπάρχουν και κάποια εναλλακτικά ψηφίσματα, αλλά το βασικό μήνυμα είναι ότι το Κοινοβούλιο θέλει στο μέλλον να έχουμε μια καλύτερη συμφωνία με το Μαρόκο και είδαμε ότι οι τωρινές ρυθμίσεις με το Μαρόκο θα πρέπει να έχουν περισσότερο βιώσιμο χαρακτήρα και οικολογικά και οικονομικά σε σχέση με την τωρινή κατάσταση. Ελπίζω ότι θα υπάρξει ευρεία πλειοψηφία υπέρ του ψηφίσματο και η συνάδελφο Κάρον Φράγκο φαντάζομαι θα επανέλθει επί του θέματο. Όσον αφορά την έκθεσή μου που αφορά το ίδιο θέμα, Πρέπει να πω ότι αυτό είναι ένα θέμα που το συζητάμε στην Επιτροπή Αλίας για μεγάλο χρονικό διάστημα και θέλω να σας εξηγήσω γιατί ε, παρότι αναφέρεται ότι δεν είναι καλές ε, οι τρέχουσες συνθήκες ε, σας προτείνω να ψηφίσουμε κατά τη έκθεση. Πρέπει να σας πω ότι η δική μου εισήγηση προς την Επιτροπή Ελία ήταν να μην συμφωνήσουμε, με, να μην εγκρίνουμε την Αλληλευτική Συμφωνία και οι λόγοι εξηγούνται μέσα στο ψήφισμα. Αυτή η συμφωνία αλληλευτικής σύμπραξης ε, θα πρέπει να θεωρείται μια συμφωνία που ωφελεί και τα δύο μέρη και έχουμε ενώπιόν μας αυτό το κείμενο που δείχνει ότι αυτή η συμφωνία δεν είναι βιώσιμη κάθε άλλο. Και η έκθεση αξιολόγησης δείχνει ότι επιβαρύνονται πάρα πολύ ε, οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι περισσότερο από ότι με οποιαδήποτε άλλη αλληλευτική συμφωνία. Η απόδοση από τη συμφωνία αυτή στην πράξη είναι αρνητική οι περισσότερε συμφωνίε αλληλευτικής συνεργασίας έχουν 40% απόδοση, ενώ αυτή η συμφωνία για κάθε ευρώ που επενδύεται έχει απόδοση 0,65 ε, ε, ευρώ, άρα είναι αρνητική για του Ευρωπαίους φορολογούμενους. Πίσω από τις συμφωνίες ελευτικής σύμπραξης ε, το σκεπτικό είναι ότι ε, αλλιεύονται τα πλεονάσματα. Δεν θέλουμε να έχουμε από θεμάτων. Άρα είναι ανησυχητικό να βλέπουμε ότι από τα 11 ε, αποθέματα τα οποία αλλιεύουμε στη συμφωνία υπάρχουν κάποια 9 από τα 11 τα οποία υπεραλλιεύονται. Επομένω, αποδεικνύεται ότι δεν αλλιεύονται τα ε, πλεονάσματα, αλλά πολύ περισσότεροι πόροι, πράγμα το οποίο αποτελεί μη βιώσιμη τακτική και πολιτική. Αυτός είναι άλλο ένα λόγος για τον οποίο ζητούμε αλλαγή. Εξηγώντα αυτά τα πράγματα λοιπόν καθίσταται σαφές ότι πρέπει ε, να περάσουμε αυτό το ψήφισμα για να αποδείξουμε και στην Επίτροπο που βρίσκεται εδώ μαζί μας ότι θα πρέπει οι συμφωνίες λαμβάνουν υπόψη όλα αυτά τα προβλήματα όπως παρατίθενται στην ε, έκθεση αξιολόγησης και θέλουμε να πούμε ότι εκ μέρους του Κοινοβουλίου δεν ήταν εύκολες οι εργασίες σε σχέση με αυτή τη συμφωνία. Ε, το Κοινοβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνενέσει με αυτέ τι συμφωνίε. Αυτή είναι μια ρύθμιση που προέκυψε από τη συνθήκη τη Λισαβόνας. Θέτει μια υποχρέωση σε εμά ω Ευρωβουλευτές να εξετάζουμε αυτέ τι συμφωνίε. Εξετάζοντα λοιπόν αυτή τη συμφωνία και με βάση αυτά τα οποία είπαν οι δύο επιτροπές που γνωμοδότησαν για αυτή τη συμφωνία, είναι σαφές ότι δεν πρέπει να δεχθούμε τις τρέχουσες ρυθμίσεις και γι' αυτό πρέπει να ψηφίσουμε κατά. Η Επιτροπή Ανάπτυξη και η Επιτροπή Προπολογισμών γνωμοδότησαν για την έκθεσή μου και οι δύο επιτροπέ αυτέ μα συνιστούν να μην εγκρίνουμε τι συμφωνίε. Αυτό είναι ένα ισχυρό μήνυμα από τι Επιτροπέ Ανάπτυξη και Προπολογισμών. Στην Επιτροπή Αλληλεία ήταν δύσκολη η ψηφοφορία και κατέληξε η Επιτροπή Αλληλεία σε θετική ψήφο υπέρ τη έκθεση και την Τετάρτη που θα ψηφίσουμε για αυτό το θέμα σίγουρα θα είναι πολύ δύσκολη η ψηφοφορία. Σας καλώ να αναλάβετε την ευθύνη την οποία μας αναθέτει η συνθήκη της Λισαβόνας και να εξετάσουμε πολύ προσεκτικά τις τρέχουσες ρυθμίσεις. δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ω εχθρική κίνηση προ του εταίρου μα προ το Μαρόκο. Επομένω, δεν είναι κάτι το οποίο συνηγορεί υπέρ ε, ε, μη σύναψη αλληλευτικών συμφωνιών με το Μαρόκο στο μέλλον, αλλά πρέπει να εξετάσουμε του όρου αυτή τη συμφωνία. Σα ευχαριστώ πολύ. Ξέρω ότι δεν συμφωνούμε όλοι οι συνάδελφοι, αλλά σα ευχαριστώ για τον επικοδομητικό διάλογο και παρόλε τι διαφορέ απόψεων ε, που, είχαμε, είχαμε γόνιμη συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε συνάδελφε. Η κυρία Κάρμεν Φράγκα Εστέδες. Είναι συνεισηγήτρια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σήμερα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση για την οποία έχει παραταθεί αυτή η ελληνική συμφωνία με το Μάρακο και αυτό σημαίνει διότι δεν ετήρησε την υποχρεωσή της να ζητήσει ε, εντολή για η Κομισιόν, ούτε επίση ε, προέβη στην συμφωνία που θα έπρεπε. Όμω δεν έχει καμία ευθύνη, δεν φταίει γι' αυτό το λόγο ο λευκός τόλο δεν να πληρώσει την ύφη. Γι' αυτό και επομένω αυτό το οποίο θέλουμε είναι να δοθεί μια λύση και θα πρέπει επομένω να αποφανθούμε θετικά. Επίση δεν συμφωνώ με αυτού οι οποίοι ε, έχουν ενστάσεις λόγω Δυτικής Σαχάρας ε, ή επί της ουσίας της αξιολόγησης και οπότε πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι ήδη από το 2006 στην ετολική έκθεση ε, της τότε Ελληνικής Συμφωνίας στο Κοινοβούλιο ε, είχε αποφανθεί ομόφωνα όσον ε, αφορά το πόσο ωφελεί το λαό της Δυτικής Σαχαράς του Σαχράου αυτή η συμφωνία διότι η, ήταν πάρα πολύ αρνητικές συνέπειες της έλλειψης συμφωνίας οπότε τα προβλήματα αυτά δεν θα λυθούν τώρα όμως εις βάρος και στις πλάτες του αλληλευτικού μας τόλου. Άρα θα πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτή τη συμφωνία και κυρία Επίτροπε βρισκόμαστε πάλι σε, στην ίδια κατάσταση ότι έχουμε ε, λιγότερο από τρεις μήνες που πρέπει να έχει κλείσει αυτό το θέμα της ε, παράτασης. Θα λήξει η παράταση που έχει δοθεί και δεν έχουμε ακόμα την, ε, την εντολή διαπραγματευτική. Όμως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την υπεύθυνη στάση του κλάδου και, του κλάδου του από Μαρόκου. Ε, γιατί έγινε σχετική συμφωνία την περσμένη εβδομάδα στι Βρυξέλλε και γι' αυτό και με τον κύριο Χάγκλουντ ε, και η φιλελεύθερη επομένω και η δική μου πολιτική ομάδα έχουμε την προφορική ερώτηση και έχουμε και αυτό το σχέδιο ψηφίσματος για να καλύψουμε το μέλλον, για να δώσουμε καινούργια θεμέλια στο μέλλον, για να μπορέσουμε να διορθώσουμε τα λάθη του παρελθόντος. Ο, και είναι επίσης κάτι στο οποίο συμφωνούν όλοι οι εμπλεκόμενοι και συμφωνώ, ελπίζω να συμφωνεί και η Κομισιόν. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Φράγκα. Σε η κυρία Δαμανάκη, πέντε λεπτά. Thank you, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί βουλευτές, καλασορίζω την ευκαιρία που μου δίνετε να μοιραστώ μαζί σας την αξιολόγησή μου ε, σε σχέση με την ε, τρέχουσα κατάσταση και τις απόψεις μου για το μέλλον της ε, αληφτικής μας συμφωνίας με το Μαρόκο. Θα ήθελα να ξεκινήσω καταρχήν με το εισαγωγικό πρωτόκολλο. Θα αποφασίσετε τώρα εάν το πρωτόκολλο αυτό μπορεί να συναυθεί ή όχι. Η Βασική Επιτροπή έχει δώσει θετική σύσταση, αλλά ξέρω ότι πολλοί από εσά δεν είσαστε πεπισμένοι. Θα ήθελα λοιπόν να σας εξηγήσω ποια είναι η θέση μας. Όπως ξέρετε, αυτό το μονοετές ε, ενδιάμεσο πρωτόκολλο συμφωνήθηκε με το Μαρόκο το Φεβρουάριο του 2011, λίγο πριν ε, εκπνεύσει το προηγούμενο. Είμαι πεπισμένη ότι αυτή η απόφαση ήταν σωστή. Ακόμα και σήμερα πιστεύω ότι κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε. Γιατί? γιατί το ενδιάμεσο πρωτόκολλο μας έδωσε το χρονικό περιθώριο να αντιμετωπίσουμε τα νομικά και πολιτικά θέματα που αφορούν την αλίευση στα ύδατα της Δυτικής Σαχάρας. Ε, πιέσαμε το Μαρόκο να μας δώσει αξιόπιστα στοιχεία και να μας πει ότι ο τοπικός πληθυσμός επωφελείται από την εκμετάλλευση αυτών των υδάτων όπως απαιτούν ε, και οι διεθνείς συμφωνίες και το διεθνές δίκαιο. Αυτές οι προσπάθειες έχουν δώσει κάποια δυνητικά θετικά αποτελέσματα. Για πρώτη φορά το τρέχον πρωτόκολλο περιλαμβάνει μια τυπική απέτηση από το Μαρόκο να μιλάει για τα ωφέλη και την γεωγραφική κατανομή τους και με αυτόν τον τρόπο ε, δημιουργείται ένα σημαντικό ε, προηγούμενο για οποιοδήποτε μελλοντικό πρωτόκολλο. Σε ό,τι αφορά τώρα τα οικονομικά και ε, περιβαλλοντικά θέματα, η εντολή για επέκταση του προηγούμενου πρωτοκόλλου δεν μας άφησε πολύ μεγάλο περιθώριο διαπραγματευτικό στις τελευταίες διαπραγματεύσεις. Δηλαδή δεν είχαμε τη δυνατότητα ουσιαστικά να συνάψουμε καλύτερη συμφωνία σε ό,τι αφορά τα οικονομικά και περιβαλλοντικά θέματα. Παρ' όλα αυτά, είναι σαφές ότι οποιαδήποτε μελλοντική διαπραγμάτευση θα πρέπει να είναι να οδηγήσει σε μια καλύτερη συμφωνία. Στο κάτω-κάτω αυτό το ενδιάμεσο πρωτόκολλο μας έδωσε τη δυνατότητα να συνεχίσουμε τις αλληλευτικές μας προσπάθειες χωρίς να υπάρξει διακοπή. Ξέρω ότι πολλοί από εσά δεν είσαστε επιπισμένοι για το αποτέλεσμα, αλλά θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό για κάποιες εκατοντάδες αλληλευτικά ευρωπαϊκά σκάφη που ψαρεύουν εκεί και κυρίως σκάφη μικρής κλίμακας, αλίας μικρής κλίμακας. Με βάση την απόφαση που πήρε το Συμβούλιο τον Ιούλιο, το πρωτόκολλο τώρα ισχύει προσωρινά. Και δεν έχουν μείνει ούτε τρίτη μήνες πριν εκπνεύσει, για να εκπνεύσει δηλαδή, γιατί εκπνέει στα τέλη Φεβρουαρίου του 2012. Ο κύριος και ε, η κυρία Φράγκα, ε, οι συγητές σας δηλαδή και πολλοί από εσά δεν είσαστε ικανοποιημένοι που αναγκάζετε το Κοινοβούλιο να πάρει θέση μόνο τώρα. Αλλά δεν είναι δικό μας λάθος. Εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να επιταχύνουμε τις διαδικασίες. Ούτω ή άλλω είμαι ικανοποιημένη που το Κοινοβούλιο ε, προέβη σε αυτή την ψηφοφορία χωρί καθυστερήσεις, σε αυτή την ολομέλεια δηλαδή, και θα γίνει μάλλον αυτό σε αυτήν την Ολομέλεια και το αποτέλεσμα θα είναι πολύ σημαντικό για όλου μα. Ούτω ή άλλω θα σεβαστούμε την ψήφο του Κοινοβουλίου. Αυτό θα ήθελα να το ξεκαθαρίσω. Η ψήφο σα την επόμενη Τετάρτη θα ληφθεί υπόψη, θα τη σεβαστούμε. Σα διαβεβαιώ επίση ότι θα λάβουμε υπόψη τι ε, συστάσει τη έκθεση Χάγκλουντ ε, και όλα τα θέματα που θέτει, καθώς και τα θέματα που αναφέρονται στο, στην πρόταση ψηφίσματος. Σε περίπτωση νέας συμφωνίας, λοιπόν, θα πρέπει να βελτιώσουμε σημαντικά το κείμενο σε ό,τι αφορά τα περιβαλλοντικά, οικονομικά και νομικά και πολιτικά θέματα. Θα ήθελα να πω τώρα δύο λόγια για τις πρόσφατες εξελίξεις στο Μαρόκο και για τις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μαρόκου. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ε, λαμβάνεται η δική σας απόφαση σήμερα, ούτως ή άλλως. Η αλλαγή που υπάρχουν στην ε, Νότια Μεσόγειο και σε κάποιες άλλες χώρες πέραν της Νότιας Μεσογείου ε, άγγιξαν και το Μαρόκο. Ποια είναι η αξιολόγηση της Κομισιόν. Η αξιολόγησή μας είναι ότι οι αρχές του Μαλόκου έχουν ξεκινήσει μια σημαντική διαδικασία μεταρρυθμίσεων Υπάρχει ε, η προσπάθεια εκπόνησης νέου συντάγματος, μεγαλύτερη δημοκρατική διαφάνεια, σεβασμός ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ε, καθώς και σοβαρές ε, βουλευτικές εκλογές που έφεραν νέες δυνάμεις στην εξουσία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλα τα επίπεδα καλωσορίζει αυτές τις αλλαγές. Ο οίκος σας ζήτησε επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση να υποστηρίξει την διαδικασία δημοκρατικής αλλαγής στο Μαρόκο. Αυτό το πλαίσιο το ξεχνάμε για να πάρουμε την αποφασή μας και ενόψει των αποφάσεών μας. Τον περασμένο μήνα η Επιτροπή Αλίας, το είπαμε στην Επιτροπή Αλίας, ότι εμείς ετοιμάζουμε την πρόταση που υποβάλλουμε στο Συμβούλιο για μια νέα διαπραγματευτική εντολή. Καταρχάς είχαμε σκεφτεί να περιμένουμε τη δική σας ψήφο της Τετάρτης, αλλά τελικά καταλάβαμε ότι θα ήταν πολύ αργά για τις εργασίες μας, ε, να το κάνουμε αυτό και ούτως ή δεν μπορούσατε να μπείτε εσείς στην ουσία. Γι' αυτό λοιπόν ε, πήραμε αυτή την πρωτοβουλία για να είμαστε έτοιμοι εγκαίρως σε περίπτωση που εσείς το Κοινοβούλιο μας δώσετε την Δετάρτη ε, θετικό μήνυμα και μας πείτε, δίνοντάς μα το πράσινο φως προχωρήστε. Κάναμε λοιπόν την προετοιμασία σε περίπτωση που εσείς θα δώσετε τη συνένεσή σας σε αυτό το πρωτόκολλο. Ποιε είναι οι βασικές παράμετροι αυτή τη καλύτερη συμφωνία με, το, με το Μαρόκο που θα πρέπει να επιδιώκουμε. Καταρχά, οικονομική κερδοφορία. Θέλουμε να επενδύουμε λεφτά, αλλά να αξίζει τον κόπο. Θα πρέπει το πρωτόκολλο αυτό να εξασφαλίζει καλύτερη χρήση των αλληλευτικών δυνατοτήτων, καθώς και συνολικά ένα καλύτερο οικονομικό ποσό που έχει αγοραία αξία, όπως είπαν και διάφορες κοινοβουλευτικές επιτροπές. Δεύτερον, για τα, την περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Αυτό τι σημαίνει. Οι αλληλευτικές δυνατότητες θα βασιστούν στις καλύτερες δυνατές ε, επιστημονικές συμβουλές και μόνο στα πλεονάσματα. Για την νομιμότητα, σε ό,τι αφορά τα ύδατα της Δυτικής Σαχάρας, θα σεβαστούμε πλήρως το διεθνές δίκαιο. Υπάρχουν διάφορες εναλλακτικές λύσεις για το πώς θα πετύχουμε κάτι τέτοιο. Εξετάζουμε όλες τις εναλλακτικές λύσεις και αν συμπεριλάβουμε και τα ύδατα της Δυτικής Σαχάρας τελικά, θα πρέπει να καταδείξουμε μέσω αυτής ενός αυστηρού μηχανισμού λογοδοσίας ότι υπάρχουν οικονομικά ωφέλη για την περιοχή και τον τοπικό πληθυσμό. Αυτό θα είναι προϋπόθεση ε, στο νέο πρωτόκολλο. Για όλα αυτά τα θέματα θα βασιστούμε στα αποτελέσματα του προηγούμενου πρωτοκόλλου, αλλά θα βασιστούμε και στις συζητήσεις ε, του Κοινοβουλίου. Το περασμένο μήνα η Επιτροπή Αλίας ζήτησε ε, να συνενέσει το Κοινοβούλιο για το πρωτόκολλο και αν τελικά συμφωνήσετε θα είμαστε έτοιμοι να κινηθούμε προς ένα καλύτερο πρωτόκολλο εν ώψη, καλύτερο πρωτόκολλο της συμφωνίας αυτής με το Μαρόκο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε Επίτροπε. Συνάδελφος ε, Λόβιν από την Επιτροπή Ανάπτυξης. Δυόμιση λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, στο μέσο της Σαχάρας ε, το Μαρόκο δημιούργησε ένα τείχος 270 ε, χιλιόμετρων, το μεγαλύτερο τείχος μετά το συνικό τείχος, το οποίο φυλάσσεται από 120.000 στρατιώτες και πάρα πολλές ε, νάρκες. Επίσης υπάρχουν και οι μάντες που μεταφέρουν άλλα τα φωσφόρου από αυτή την περιοχή. Από το 1975 με βόμβες ε, Ναπάλ και Φωσφόρου το Μαρόκο κατέλαβε ε, την ε, Δυτική Σαχάρα και αυτό αποτελεί έγκλημα στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου. Η αλληλευτική συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μαρόκου που συμπεριλαμβάνει τα ύδατα της Δυτικής Σαχάρας είναι παράνομη. Αυτό έχει εκφραστεί ως πόρισμα από την νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου με βάση προηγούμενη απόφαση και της Επιτροπής θα έπρεπε να καθορίσουν αν αλλιεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Δυτική Σαχάρα και δεύτερον εάν το οικονομικό αντιστάθμισμα ωφελούσε το λαό της Δυτικής Σαχάρας και αν αυτό γινόταν με συνένεση του λαού της Δυτικής Σαχάρας. Τώρα υπάρχουν οι απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα. Το 74% του στόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλιεύει στα ύδατα της Δυτικής Σαχάρας και ο λαός αυτής της περιοχής δεν έχει δώσει τη γνώμη του για αυτό το θέμα. Αγαπητοί συνάδελφοι, τις απαντήσεις που έδωσε το Μαρόκο στην Επιτροπή πριν από ένα χρόνο για τα ερωτήματα αυτά τις είδα. Και είναι 100% ξεκαθαρό ότι το Μαρόκο δεν ε, θα αναγνωρίσει ότι υπάρχει Δυτική Σαχάρα. Δεν αναφέρουν ποτέ τη Δυτική Σαχάρα. Και καθίσατε σαφέ και κάτι ακόμη, ότι το Μαρόκο δεν χρειάζεται αυτή τη συμφωνία. Το Μαρόκο έχει ένα εγχώριο στόλο, μεγαλύτερο από το στόλο τη Ισπανία. Και ο στόχο του είναι να τριπλασιάσουν ε, τη συμβολή τη αλληλεία στο ΑΕΠ, να διπλασιάσουν ε, την ε, απασχόληση στον τομέα τη αλλήλία, καθώ και τα αλλιεύματα. Και για αυτού του λόγου δέχθηκε τη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση το 1999 το Μαρόκο. Είναι ξεκάθαρο ότι το Μαρόκο θέλει να κρατήσει την, Ευρωπα... συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο και μόνο για ένα λόγο. Για να νομιμοποιήσει ε, την κατοχή τη Δυτική Σαχάρα, κάνοντα συνένοχο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πραγματικά θα είναι όνειδο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση αν εμεί ω υπέρμαχοι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη Διεθνού Δικαιοσύνη και Δημοκρατία ε, συνενέσουμε σε αυτή την επονίδηση τη συμφωνία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τη συνάδελφο Λέβιν. Συνάδελφο Αλφόνση, Επιτροπή Προπολογισμών. Ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Η Επιτροπή Προπολογισμών ήθελε να μην εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την Συμφωνία αυτή Ευρωπαϊκή Ένωση και Βασιλείου του Μαρόκου. Θέλω να τονίσω ότι αυτή η άρνηση ε, δεν θα έχει πρακτική συνέπεια, γιατί αυτή η συμφωνία ε, συνέβη τον Φεβρουάριο του 2011 και εκπνέει σε ένα μήνα δηλαδή. Ουσιαστικά η Επιτροπή Προπολογισμών αρνήθηκε και μια πρόταση που ήθελε να, ε, για να μην δεχτεί την δέσμευση για τον προπολογισμό. Θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα ουσιαστικά για τις αρνητικές συνέπειες σε περιβαλλοντικό επίπεδο. Γιατί υπάρχει υπεραλίευση σε αυτά τα ύδατα και σε ό,τι αφορά τις δαπάνες ε, υπάρχει, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα τα ύδατα αυτά, ε, τα τρία τέταρτα των υδάτων ουσιαστικά συνδέονται με την Δυτική Σαχάρα. Αν ε, το, το Κοινοβούλιο δεχθείτε αυτό που λέμε εμείς, θα είναι ένα ισχυρό μήνυμα για τις μελλοντικέ διαπραγματεύσεις και ένα ισχυρό μήνυμα για την κυβέρνηση του Μαρόκου, όπου τη στιγμή όπου σε όλη την Μεσόγειο υπάρχει ένας αέρας δημοκρατίας, ε, θα πρέπει να, να πνέει ο ίδιος αέρας και για το λαό της Σαχάρας. Ευχαριστούμε τον συνάδελφο Αλφασίν. Ο μιλητέ εκ μέρου των πολιτικών ομάδων, συνάδελφο Κάντετ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα καταρχήν να μιλήσω για το ενδιάμεσο πρωτόκολλο. Ω και ο εκ μέρου τη ομάδα μου, θα ήθελα να εκφράσω το ένα μήνυμα προ τον εισηγητή. Ελπίζω ότι στην έκθεση για τη χρηματοδότηση των ελευθερικών πόρων και τη αλληλεία, όπου είναι σκιώδη συγκητή ο κ. Χάγκλουν και εγώ είμαι εισηγητή, θα μπορέσουμε να συζητήσουμε λεπτομερέστερα για την έκθεση αυτή. Και υπενθυμίζω ότι πάντοτε ήμουν ανοιχτό σε συζήτηση για όλα τα θέματα, πάντοτε όποτε δουλεύαμε και θα δουλεύουμε μαζί θα είμαι ανοιχτό. Η συμφωνία ε, μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μαρόκου είναι παράταση κατά ένα έτος μιας προηγούμενης συμφωνίας. Αυτό μας προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτή η συμφωνία λήγει στις 27 Φεβρουαρίου του 2012, δηλαδή σε δύο μήνες, όπως είπε και ο κύριος Αλφωσίν προηγουμένως. Επιτρέπει σε 10 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αλλιεύουν στα ύδατα του Μαρόκου και να ωφελείται από αυτό ο τοπικός πληθυσμός σε όλη την επικράτεια του Μαρόκου μπορούν να λεύουν τα σκάφη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπενθυμίζω ότι ψήφισαν οι συνάδελφοι υπέρ αυτή τη έκθεση, διότι είναι προ αμοιβαίο όφελο. Η έγκριση αυτή της συμφωνίας θα επιτρέψει διαπραγματεύσει για μια νέα συμφωνία αλληλεία με νέα κριτήρια. Αν απορρίψουμε αυτή τη συμφωνία θα δώσουμε ένα πολύ αρνητικό μήνυμα για όλη αυτή την περιοχή και μάλιστα σε μια περίοδο εκδημοκρατισμού. Το Μαρόκο είναι απαραίτητο εταίρο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και η υποστήριξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν περνάει μόνο μέσω διακηρύξεων που έχουμε πολλέ. αλλά και και μέσω συγκεκριμένων δράσεων. Η ομάδα μου και η ομάδα των φιλελευθέρων ε, δίνει ένα ισχυρό σήμα προς την Επιτροπή για μια συμφωνία που θα είναι και αποδοτική και οικολογικά βιώσιμη και θα επιτρέπει σωστή χρήση των αλληλευτικών δυνατοτήτων για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας υπενθυμίζω όμως ότι θα πρέπει καταρχήν να έχουμε ψηφίσει το ενδιάμεσο πρωτόκολλο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Κάντεκ συνάδελφος ρόντου, για δύο λεπτά και πάλι. Ε, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Επίτροπε, η Συμφωνία Αλίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μαρόκου απασχολεί το Κοινοβούλιο εδώ και πάνω από ένα χρόνο. Και είμαι βεβαία ότι μετά την ε, αυριανή ψηφοφορία θα συνεχίσει να μας απασχολεί. Αυτό το θέμα ε, μας έχει κινητοποιήσει και το συζητάμε σε όλο το Κοινοβούλιο και όλες οι πολιτικές ομάδες, τις τελευταίες ομάδες και τις τελευταίες εβδομάδες συζητούν ε, ε, με αντιφατικά επιχειρήματα αυτή τη συμφωνία. Θα πρέπει να δούμε ποια είναι η ανάλυση αυτής της έκθεσης. Εμείς ε, στην, συμφωνία, στην Επιτροπή Αλίας είδαμε ότι δεν είναι βιώσιμη οικολογικά αυτή η συμφωνία διότι οδηγεί σε υπεραλίευση. Στην, ε, στις συζητήσεις μέχρι τώρα δεν έχει τονιστεί αρκετά αλλά είναι ένα βασικό σημείο είναι καταστροφική η κατάσταση των υδάτων των θαλασσών παγκοσμίω και δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να υπεραλλιεύει σε ξένα ύδατα, αλλά και από οικονομική πτυχή δεν είναι ενδιαφέρουσα, δεν είναι συμφέρουσα αυτή η συμφωνία. Επιπλέον υπάρχει και το θέμα της Δυτικής Σαχάρας. Είμαι βεβαία ότι όλοι μας συμφωνούμε ότι η συμφωνία αυτή θα πρέπει να ισχύει μόνο σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Δεν υπάρχει συμφωνία όμως του λαού της περιοχής. Το ότι στο μέλλον θα αλλάξουν όλα μπορεί να είναι ένας παράγων παρηγοριάς, είναι μια ελπίδα και ελπίζω ότι με την πρότασή μας θα δώσουμε στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο δυνατότητα να κάνουν σωστές συμφωνίες στο μέλλον. Ο μοναδικό λόγο που μπορούμε να ψηφίσουμε υπέρ είναι ότι είμαστε λίγο πριν τη λήξη του πρωτοκόλου και δεν θέλουμε να διακόψουμε την ισχύουσα κατάσταση και να επιβαρύνουμε τι διαπραγματεύσει για τη νέα συμφωνία. Όλε οι προσπάθειε μα ελπίζουμε ότι θα ευωθούν στο νέο πρωτόκολλο. Είναι κάτι το οποίο προσδοκώ και μάλιστα το περιμένουμε και με δέσμευση όλων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τη συνάδελφό Ρόντου, συνάδελφο Ντέιβι, ένα μισή λεπτό. Χωρίς μικρόφωνο. Ορισμένοι από εμά ε, αισθανόμαστε οργή όσον αφορά την ισχύουσα συμφωνία. Ρίξτε μια μαριά όσον αφορά την μελέτη αξιολόγηση και θα μπορέσετε να διακρίνετε πού πάσχει αυτή η συμφωνία. Πρόκειται για μια μελέτη η οποία ξεκαθαρίζει ότι πρόκειται για την οίκιστα επιτυχημένη από όλε τι συμφωνίε που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για μια συμφωνία στην οποία 36 εκατομμύρια ευρώ τα βάζουν την τσέπη του φορολογούμενοι και τι έχουμε σε αντάλλαγμα <clears throat> τα, τα ψάρια που πιάνουν δεν έρχονται εδώ, πάνε αλλού, πάνε στην Αφρική, πάνε στην Ασία. Οι δε πλειοκτήτες, πρόκειται για 80 κριτικά σκάφη, οι οποίοι τι, βάζουν, βάζουν 2 εκατομμύρια, δεκάρες Οπότε, ε, τι γίνεται με το θέμα της βιωσιμότητας δε. Βλέπουμε ότι αλλιεύουν σε υδατά τα οποία μάλλον υπερ αλλιεύονται. Άρα πέφτει και η υπόθεση τη βιωσιμότητα. άρα. Ε, κάντε ό,τι μπορείτε παρακαλώ κύριε Επίτροπε να, να κάνετε μια διαπραγμάτευση που πραγματικά να καλύπτει τα κοινωνικά κριτήρια και τι ε, βιωσιμότητε. αυτά τα οποία αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση, στην ε, διακήρυξη κλπ. Όχι, όχι, δεν φταίτε εσεί για εκείνη την τραγική ρύθμιση η οποία ισχύει σήμερα. Ευχαριστούμε κύριε Ντέβις. η ρουέβα Ιρουέβα, μισή λεπτό. Σας ευχαριστώ. Βεβαίω. Είναι αυτονόητο ότι εγώ όχι μόνο δεν θέλω να παραταθεί ισχύω συμφωνία, αλλά και είμαι κατά και μια νέα συμφωνία. Και αυτό διότι έχουμε, ε, έχουμε τώρα θέματα νομικά, οικολογικά και ε, οικονομικά. Γιατί μιλάει και διαπραγματεύεται το Μαρόκο ε, ε, για, για, για κάποιου ελευθερού πόρου που δεν τους ανήκουν. Πρόκειται εδώ πέρα για το ότι αφήνει έξω από το πλαίσιο των έξω από την εικόνα, από το οποίο του Σαχράουι. Και θέλουν επομένω τώρα ε, να καλυφθούν και οι επιθυμίες αλλά και τα συμφέροντα του τοπικού πληθυσμού. Όμως, όμως αυτό παρά το ότι είναι αίτημα γενικό κανεί δεν το έχει λάβει υπόψη. Η προηγούμενη συμφωνία ήταν μια τραγωδία γιατί με τίποτα δεν επέφερε κάποιο είδους ε, κάποιο του κέρδη, το αντίθετο ε, ήταν μια διασπάθηση των ε, πόρων και επομένως όσον αφορά τις συμφωνίες είχαμε πει ότι θα πρέπει να γίνεται αλίευση εκεί που υπάρχει κάποιο είδους ε, πλεόνασμα. Όμως σε αυτή την περίπτωση βρισκόμαστε σε φάση, σε κατάσταση, σε περίπτωση υπεραλίευσης από τους τοπικούς και οπότε τώρα τι κάνουμε, ερχόμαστε και προσθέτουμε εκεί πέρα και τους Ευρωπαίους. Άρα είπαμε λοιπόν έχουμε τρεις λόγους να πούμε κατά ε, νομικά, οικολογικά, ε, οικονομικά. Γι' αυτό και θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να καμφθεί το Κοινοβούλιο ε, από τις πιέσεις της κυβέρνησης του Μαρόκου γιατί εδώ πέρα διακυβεύεται η εξοπιστία μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Ρωμέβα Ιρουέδα. Για μισή λεπτά συνάδελφος Φερέιρα. Ευχαριστώ πρόεδρε κύριε Επίτροπε. Με αυτή την πρόταση παράτασης αυτής της συμφωνίας, η Κομισιόν έπεσε σε μια αντίφαση και διέπραξε ένα λάθος. Ζήτησε από εξωτερικούς σύμβουλους να κάνουν μια εξπόστ αξιολόγηση για τις τέσσερα, τα τέσσερα χρόνια που κράτησε η συμφωνία. Νομίζω ότι και από οικονομικής πλευράς και από άποψη χρησιμότητας τη συμφωνία για τον αλληλευτικό μα κτόλο, αλλά και από οικολογική πλευρά, ήταν αρνητική αυτή η συμφωνία. Δεδομένου του ότι τα διάφορα αλλιεύματα είναι σε ολένα και χειρότερη κατάσταση. Επιπλέον, η Κομισιόν ε, μπροστά σε αυτή την έκθεση μας λέει Μα αυτή η έκθεση δεν εκφράζει την άποψη της Κομισιόν. Αλλά όμως εσείς δεν έχετε κάποιον αντίλογο σε αυτά τα στοιχεία. Δεν έχετε κάτι να αντιτάξετε. Ο λόγος για τον οποίο ήταν, ήμασταν αντίθετοι το 2005 και για τον οποίο πάλι θα είμαστε αντίθετοι τώρα σε αυτή τη συμφωνία είναι ότι ουσιαστικά δεν σεβόμαστε το διεθνές δίκαιο έτσι. Η συμφωνία αυτή προβλέπει ε, την εκμετάλλευση κάποιων φυσικών πόρων ε, επί των οποίων δεν έχει κυριαρχεί ουσιαστικά το Μαρόκο. Από το 1975 υπάρχει απόφαση του Διεθνούς ε, Δικαστηρίου ε, και ποτέ δεν έχει ε, αποφασιστεί ότι το Μαρόκο έχει κυριαρχία πάνω στα ύδατα της Δυτικής Σαχάρας. Επίσης υπάρχει και το ψήφισμα του 2009 για τις οικονομικές δραστηριότητες και άλλες δραστηριότητες που αφορούν τον τόπιο πληθυσμό που δεν είναι αυτόνομος. Ο πληθυσμός της Σαχάρας ποτέ δεν μπόρεσε να πει την άποψή του καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής τον έχουμε αγνοήσει. Αντίθετα από αυτά που λέτε, κύριε Επίτροπε, πρέπει να τον ακούσουμε. Γιατί ουσιαστικά αλλιώ αγνοούμε το διεθνέ δίκαιο. Δεν πρέπει να ακούμε μόνο τι λέει το Μαρόκο, που λέει ότι επωφελείται και ο πληθυσμό τη Σαχάρα. Εμεί δεν έχουμε πρόβλημα να συνάπτουμε συμφωνίε με τρίτε χώρε, αλληλευτικέ συμφωνίε. Αντίθετα, έχουμε υποστηρίξει πάρα πολλέ ε, συμφωνίε παρά τα προβλήματά του. Αλλά τα, οι συμφωνίε αυτέ θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα τη ελεύθερη έκφραση των κυρίαρχων λαών. Και δεν θα πρέπει να λαιλατούμε ουσιαστικά, γιατί αυτό κάνουμε, λαιλατούμε του φυσικού πόρου, ε, μαζί με το Μαρόκο. Είμαστε συνένοχοι του Μαρόκου ουσιαστικά θα έπρεπε ουσιαστικά να αποκλείσουμε τα ύδατα της δυτική Σαχάρας και να ξεκινήσουμε έναν ε, πραγματικό διάλογο με τον τόπιο πληθυσμό. Το Μαρόκο ε, κατέχει τη Δυτική Σαχάρα από τη δεκαετία του 1970 και αν αυτή η αλληλευτική συμφωνία προχωρήσει, τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παραβιάζει το διεθνέ δίκαιο. Το ξέρει αυτό το Γενοβουλίο, το ξέρει αυτό η νομική πτώση Συμβουλίου. Και αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε από πλευρά του Μαρόκου είναι 36 εκατομμύρια το οποίο θα πληρώνει αυτή η χώρα κάθε χρόνο. Και οπότε αυτό θα είναι λαιλασία των αλληλευτικών πόρων. Εμεί έχουμε διαβεβαιώσει του Σαχράου ότι θα ωφεληθούν από την εν λόγω αλληλευτική συμφωνία, όμω δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι τελικά θα του καταπιεί, θα του καπελώσει το Μαρόκο. Όμω παρόλα αυτά η Κομισιόν δεν δίνει δεκά Άρα για το deal αυτό. Βέβαια, οι, τα δικά μας σκάφη πηγαίνουν εκεί και φροντίζουμε ώστε να ωφεληθούν το πηγή. Θα ήταν κρίμα να σταματούσε αυτή η πρακτική. Οπότε αυτό δείχνει ότι δεν έχει κανένα έλεγχο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά ε, την ελευθερική μα δημοκρατία. Τώρα, οι Lib Dem, οι φιλελεύθεροι στην Αγγλία, προσπαθούν κάτι να κάνουν, έχουν υποβάλει ένα ψήφισμα και θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να κλείσει αυτή τη συμφωνία όσο γίνεται πιο σύντομα. Και αυτό σα δείχνει πόσο λίγο νοιάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν του χαίρεται καρφί ότι γίνεται σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε, κύριε Άγνιου. Ο συνάδελφο Ντέβι έχει μια ερώτηση συμπληρωματική. Ντέβι, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τον αξιότιμο συνάδελφο. Τι στοιχεία έχει ότι οι φιλελεύθεροι δημοκράτε του κύριου Χάγκλαντ προσπάθησαν να ματιώσουν αυτή τη συζήτηση. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι αναλυθέ. Ο προλαλής χωρί μικρό. Πρόεδρε, πρόεδρε, οι συντονιστέ θέλανε να αφαιρέσουν την ψήφο το οποίο δεν, δεν είναι και πολύ δημοκρατικό. Θα μα καπελώσουν. Ευχαριστούμε συνάδελφοι. Αυτέ ήταν οι παρεμβάσει εκ μέρου των πολιτικών ομάδων και ακολουθούν οι συνάδελφοι. Συνάδελφο Πατρέων Εύε, δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, Κυρία Επίτροπε, η εξωτερική διάσταση τη ε, κοινή ελευθερική πολιτική, αλλά και αυτέ οι συμφωνίε ελευθερικέ με τρίτε χώρε αποτελούν ένα στοιχείο απαραίτητο για την κοινή ελευθερική μα πολιτική. Έχουμε αυτή την ελευθερική συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση Μαρόκου που είναι πάρα πολύ σημαντική όσον αφορά την Νότια Ευρώπη σε μια τέτοια πολιτική συγκυρία κατά την οποία είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην κλεινόμαστε στον εαυτό μα. γιατί έχουμε αυτέ τι συμφωνίε συνεργασία, οι οποίε ε, δίνουν την ευκαιρία στον κοινοτικό ελευθερικό στόλο ούτω ώστε σε κάποιο τέτοιου είδου ε, επικράτεια να μπορούν να ασκήσουν τα δραστηριότητά του και έτσι θα έχουμε κάποια σημαντική παραγωγή, ούτω ώστε να τροφοδοτείται η αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, επίση, πρόκειται για ένα σημαντικό ρόλο τον οποίο θα παίξουμε στην οικονομική σκηνή των άλλων χωρών. Θα τι βοηθήσουμε και αυτέ να αναπτυχθούν και να αναπτυχθούν και κοινωνικά, γιατί έχει αναφερθεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση με την δραστηριότητα τη αυτή θα πρέπει να είναι ε, ε, σύντονη, θα πρέπει να είναι συνεπή με τι διεθνεί τη δεσμεύσεις και όσον αφορά την ε, διατήρηση, την προστασία του περιβάλλοντος, του ελευτικού πόρου και γι' αυτό, εάν έχουμε μια τέτοια βιωσιμότητα στη δραστηριότητα αυτή κατόπιν συμφωνία, αυτό θα βγει σε μια διαχείριση βιώσιμη στους ελευτικούς πόρου και αυτό θα γίνει μέσω αυτής της ρήτρα διαφάνειας. Και έτσι θα προστατευθούν οι ελευτικοί πόροι όσον αφορά την ε, λίευση από τα σκάφη μας σε τρίτες χώρες και... Ε, αυτό θα αφορά μια νέα συμφωνία. Μια συμφωνία που θα πρέπει να διέπεται από κάποιο είδους αξιόπιστα επιστημονικά στοιχεία και θα πρέπει επίσης να την χάνει εποπτείας, παρακολούθησης όσον αφορά την εφαρμογή της. Αυτό αφορά και τα οικοσυστήματα, αυτό αφορά και τους εμπλεκόμενους άλλους όπως τους τοπικούς πληθυσμούς. Δυστυχώς θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει τηρήσει το ότι δεν, έχει, δεν, έχει, δεν κάνει μάλλον αυτό, δεν κάνουν οι άλλοι αυτό που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά αυτά τα ίδια ύδατα. Ευχαριστούμε. Συνάδελφος Μιλάνα, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε η χειρότερη συμφωνία, η χειρότερη παράταση, το χειρότερο αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά τις προσπάθειες των τελευταίων χρόνων. Αυτή είναι η κατάληξη της ε, συζήτησης. Δεν πρέπει να αρχιοθετήσουμε όλη αυτή η συζήτηση. Αν η Επίτροπος περισσότερο από την ε, Κομισιόν μας ζητάει να εγκρίνουμε αυτή τη συμφωνία, τότε θα πρέπει να σκεφτούμε κάτι εντελώς καινούριο, να δούμε τι μπορεί να συμβεί τα επόμενα χρόνια. Δεν νομίζω ότι οποιοδήποτε όπως εγώ είναι υπέρ του, του λαού της Δυτικής Σαχάρας μπορεί να υποστηρίξει μια τέτοια συμφωνία. Δεν μπορούμε εμείς να υποκαταστήσουμε τώρα Ε, δεν μπορούμε να, να βρούμε εμείς λύση, δεν μπορούμε να είμαστε εμείς οι σωτήρες. Ε, είναι μια είναι ένα πρόβλημα ανάμεσα στη Δυτική Σαχάρα και στο Μαρόκο που κρατάει 30 χρόνια. Δεν μπορούμε να βρούμε εμείς ε, λύση τη στιγμή που κανένας δεν μπόρεσε να βρει λύση, τη στιγμή που ο ΙΕ επί 30 χρόνια έχει μια αποστολή και που δεν υπάρχει λύση. Πώς θα, θα βρούμε εμείς τη λύση τώρα, ε, μέσω της αλληλευτικής συμφωνίας, τώρα. Ναι στο ψήφισμα, ναι στην παράταση της, ε, του πρωτοκόλου αλλά για να δώσουμε τη δύναμη στην Κομισιόν να δείξει στεναρή θέση, ούτω ώστε η συμφωνία αυτή να είναι να δώσει ένα σωστό μήνυμα και να είναι συμβατή με την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι δυνατόν η Βαρόνια Άστο να μην ασχολείται καθόλου με το λαό της Δυτικής Σαχάρας. Δεν είναι δυνατόν κάτι τέτοιο. Ευχαριστούμε. Συνάδελφος Βάγγελ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, επέστρεψα χθε από την, την Τούφα και είδα τι πλεονεκτήματα χάρη στις πολιτικές μας έχουν οι Σαχαράουι. Τα είδαμε τα ίδια με τα μάτια αυτά τα πλεονεκτήματα. Αυτή η συμφωνία πρέπει να την απορρίψουμε. Είμαι υπέρ της καταψήφισης αυτής της συμφωνίας για πολιτικούς, ηθικούς και διεθνείς νομικούς λόγους. Αυτή η συμφωνία δεν είναι μια κλασική, μια κοινή αλληλευτική συμφωνία. Είναι κάτι διαφορετικό. Είναι μια συμφωνία όπου τα αλληλευτικά δίκτυα, η δικαιοσύνη και το, και το δίκαιο θα μπερδευτούν όλα μαζί. Ο λαός της Δυτικής Σαχάρας χυμάζεται από την κατοχή του Μαρόκου. Γι' αυτό δεν πρέπει να επιτρέψουμε αυτή τη συμφωνία. Δεν είναι μια συμφωνία για την αληθική προσπάθεια. Πρόκειται για μια πολιτική απόφαση και αν ψηφίσουμε ναι είναι λάθος. Ευχαριστούμε τον συνάδελφο Βάιγκλ. Για ένα λεπτό, συνάδελφο Ταβάρε. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ψηφίσουμε μια συμφωνία η οποία είναι ιδιάζουσα τμήμα του στόχου αυτής της συμφωνίας ε, ε, είναι μια περιοχή ε, που αποτελεί τμήμα μιας χώρας και μιλάμε για τα αλληλευτικά αποθέματα μιας χώρας, ενός λαού, που δεν έχει δικαίωμα έκφρασης. Αντίστοιχη με την κατάσταση που είχαμε στο Ανατολικό Τιμόρ και πολύ συχνά η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, επαναλαμβάνει ε, το τι ισχύει για μια χώρα που εν μέρη είναι ε, τελή υποκατοχή. Πάντοτε το τονίζαμε αυτό στην Ινδονησία και στην Αυστραλία. Μπορούμε να αλλιεύουμε σε μια χώρα αλλιεύματα τα οποία δεν ανήκουν σε αυτή τη χώρα. Κάνουμε μια συμφωνία με το Μαρόκο για αλλιεύματα που δεν ανήκουν σε αυτή τη χώρα. Δεν μπορεί να υπάρχει συμφωνία με μια χώρα σχετικά με πόρους που δεν ανήκουν στη χώρα αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Συνάδελφε Ταβάρες, συνάδελφος Μάτο Αντροβέρ, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. Δεκέμβριο μήνα συζητάμε αυτή την συμφωνία, ή την πάση συμφωνία που θα λήξει αυτή ενίσχυση ε, σε δύο μήνε. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και, και την Ισπανία. Δεν θα πρέπει τώρα βέβαια να γίνεται αυτό μια πρόφαση για κάποιο άλλο είδου αιτήματα και διεκδικήσει. Ε, νομίζω όμως ότι η ισχύουσα συμφωνία είναι οίκιστα ικανοποιητική για πολλά. Τώρα να δούμε τι, ποιες είναι οι συνέπειες για κάποιες τρίτες χώρες ε, και να δούμε πόσο σημαντικό είναι το να γίνουν αυτές οι ρυθμίες που πρέπει για σημαντικούς μας γείτονες όπως το ε, Μαρόκο. Άρα να γίνει μια ισορροπημένη συμφωνία, να είναι δίκαιη, να ωφελεί όλους τους προσυπογράφοντες και επίσης να επιτρέπει στο αλληλευτικά μας να συνεχίσουν την επιχειρηματική δραστηριότητα. Επίσης θα πρέπει να είναι κάτι το βιώσιμο οικονομικά. Θα πρέπει να έχουμε προστασία των πόρων, αλλά θα πρέπει να έχουμε και κάποιο είδους επιπτώσεις θετικές και από εργασιακή πλευράς και οικονομικής. Οπότε θα πρέπει να είμαστε συνεπείς με τις δεσμεύσεις μας και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τη γνώμη του κλάδου. Επομένως, θα πρέπει να απαιτήσουμε και από την άλλη πλευρά να τηρηθούν τα όσα η άλλη πλευρά οφείλει στους δικούς μας αλληλείς. Επομένως, χωρίς να έχουμε καθυστερήσεις, προχωρήστε σε διαπραγματεύσεις. Οι κακές διαπραγματεύσεις οδηγούν σε κακή κατάληξη και περί τούτου έχουμε πάρα πολλές αποδείξεις. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. συνάδελφος Χάρτου. Uh, uh, θα ήθελα να ζητήσω τον uh, αγαπητό συνάδελφο ποιος θα υποφελεί το περισσότερο, όλα τα κράτη-μέλη ή μόνο η Ισπανία. Πείτε. Όπως και να τα πράγματα, εγώ θα σας πω ότι όταν ένα κράτος μέλος ωφελείται, όλοι ωφελούμεθα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ και ακολουθεί συνάδελφος Αντρές Μπαρέ, 1,5 λεπτό. Πρόεδρε, εμεί οι σοσιαλιστέ θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό να εγκριθεί αυτή η παράταση. Θα είναι κρογωνίως λήθο, ούτω ώστε να προχωρήσουμε σε μια νέα συμφωνία, διότι ε, σε τρεις μήνες εκπνέει η συμφωνία. Το προείπε η Επίτροπος και θα πρέπει να κάτσουμε για να ζυγίσουμε το πόσο αρνητικές ήταν μέχρι τώρα οι συνέπειε οικονομικής. οικονομική. Όμως επίσης δεν κάθεται να ζυγίσετε το τι γίνεται όσον αφορά ε, αυτό το οποίο μόλις τώρα ε, υπευλήθη ω ερώτηση. Έχουμε 800 εργαζομένους σε αυτέ τι 11 χώρε που έχουν δουλειά λόγω αυτή τη συμφωνία και έχουμε επίσης άλλες χιλιάδες θέσει εργασία που ωφελούνται οι Μαροκινοί, οι Σαχραούοι κλπ. Η βιωσιμότητα φυσικά και είναι σημαντική επίσης Αναφέρθηκε τι γίνεται με την έκθεση ex post. Θέλουμε για την προσεχή συμφωνία επιστημονική τεκμηρίωση γιατί έτσι θα πρέπει ε, να λάβουμε υπόψη ότι έχουμε μόνο 10% εκμετάλλευση των όσων μπορούσαμε να αλλιεύσουμε. Ε, λέγεται ότι θα πρέπει να, να βελτιώσουμε αυτήν την συμφωνία την υπάρχουσα. Επιδέχεται βελτίωση. Θα πρέπει να γίνει επί τη βάση τη ε, συμφωνία τη συνθήκη τη Λισαβόνα και θα πρέπει επίση να υπάρχει και μια έκθεση συνοδευτική που να λέει λεπτομεριακά πώ θα ισχύσει και πώ όλα αυτά συνάδουν το διεθνέ δίκαιο, διότι εμεί νομίζουμε ότι θα πρέπει όλοι να ωφελούνται και θα πρέπει η αρχιτεκτονική τη καινούργια συνθήκη να θεωρηθεί σημαντική ούτω ώστε να καλυφθεί η συμφωνία σύνδεση Μαρόκο Ευρωπαϊκή Ένωση να ληφθεί υπόψη η κοινωνική πτυχή, διεθνεί συμφωνίε, η αλληλεγγύη και το, το πόσο στρατηγική σημασία έχει το, το, το πώς θα τοποθετηθούμε στην διεθνή σκηνή με αυτή την καινούργια συμφωνία. Ευχαριστούμε τη συνάδελφο Ανδρέα Μπερέα. Τελευταίο αγορητής ο κ. Μπέρμαν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εκ μέρους του συναδέλφου Βέσλουν, θα ήθελα να διαβάσω το εξή κείμενο. Η νομική υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατέληξε στο ότι η Ελληνική Συμφωνία είναι κατά του διεθνού δικαίου, διότι το, τα Ηνωμένα Έθνη ποτέ δεν αναγνώρισαν τι απαιτήσει του Μαρόκου της τη Δυτική Σαχάρα. Δεν γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα του λαού τη Δυτική Σαχάρα και αυτή η συμφωνία δεν του συμφέρει δεν, θα έπρεπε τα ε, σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, να μην αλλιεύουν ε, στα ύδατα της Δυτικής Σαχάρας. Το τρέχον πρωτόκολλο είχε την μεγαλύτερη, το, είχε το μικρότερο δίκτυο ωφελίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με όλες τις άλλες αλληλευτικές συμφωνίες και δεν συνεισφέρει στην αύξηση των υποδομών και των δυνατών του Μαρόκου. Ευχαριστούμε τον συνάδελφο Μπέρμαν. Αν διαβάζατε λίγο πιο αργά θα ήταν ε, λίγο καλύτερα και για τους διερμηνείς, λέει ο Πρόεδρος. Είχατε χρόνο να διαβάσετε λίγο πιο αργά ε, το κείμενο που διαβάζατε για να μπορούν να το καταλάβουν και οι συνάδελφοι στις άλλες γλώσσες. Ε, ζητώ συγγνώμη από τους διερμηνείς, λέει ο, ο κύριος Μπέρμαν, γιατί του συμπαθώ και ιδιαίτερος. θεωρήστε το αυτό σχόλιο και παρατήρηση προς όλους τους συναδέλφους. Όταν έχετε κείμενα που διαβάζετε, ας τα διαβάζετε λίγο πιο αργά. Περνάμε στο Catch the Eye, συνάδελφος Νικολέσκου. Κύριε Πρόεδρε, η Αλληλευτική Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Μαρόκου δεν είναι καθόλου μια συμφωνία εταιρικής σχέσης. Όλοι οι συνάδελφοι το είπαν και δεν είναι και σωστό για την Ευρωπαϊκή Ένωση το να μην λαμβάνει υπόψη την προστασία των αλλιευμάτων, ε, το να μην λαμβάνει υπόψη τα δικαιώματα επίσης των πολιτών της περιοχής. Ήκε και η ώρα να εντατικοποιήσετε το διάλογο με τους κατοίκους, όπως και με άλλες περιοχές του κόσμου, με την Τουρκία, με, την, με περιοχές που είναι γύρω από τον Εύξηνο Πόντο κτλ. Ευχαριστούμε τον συνάδελφο Νικολέσκου, συνάδελφο Ρέγνα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ είμαι Αυστριακή, μια χώρα περίκλειστη, χωρίς πρόσβαση στη θάλασσα και εξετάζουμε την συμφωνία αυτή με το Μαρόκο όχι από ίδιο συμφέρον. Ενδιαφερόμαστε για τη βιώσιμη αλληλεία και όχι για μια αλληλεία που θα καταστρέφει τα ύδατα. Ε, αν ψηφίσουμε αυτό το πρωτόκολλο θα είναι σαν να λέμε ναι σε μια οικολογικά μη βιώσιμη συμφωνία και κάθε χρόνο κοστίζει αυτό 36 εκατομμύρια ευρώ για την Ευρωπαϊκή Ένωση κάτι το οποίο δεν ωφελεί κατά, κατά κανένα τρόπο τις θέσεις εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, η Δυτική Σαχάρα θα έπρεπε να έχει ένα δίκαιο μερίδιο τη αλληλεία για τα δικά τη παράκτια. Θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι δεν υπεραλλεύονται οι δικοί τη πόροι. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να τηρούμε εμεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σύμφωνα με τι αξίε μα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τη συνάδελφο Ρέγκνερ. Συνάδελφο Φάντσο Πρεσίντο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Λιτή Συμφωνία με το Μαρόκο ισχύει διότι έγινε παράτασή της αυτοδίκαια. Αυτό το οποίο εξέπνευσε και έληξε είναι κάποιες αντισταθμίσεις που περιέχονται σε κάποιο προσερτημένο πρωτόκολλο. Έγινε επομένως αυτή η προσωρινή παράταση και βέβαια και τον Κοινοβούλιο ήταν σύμφωνη γνώμη του, σύμφωνα με τη συνήθεια Εγώ είμαι πάντω για τι διαπραγματεύσει αυτέ υπέρ, γιατί πρώτα πρώτα θα αυτό αφορά τι σχέσει μα με το Μαρόκο. Θέλουμε να τι σφίξουμε, δεν είναι εξαίρεση ελία. Επίση, οι επιπτώσει είναι πάρα πολύ σημαντικέ όσον αφορά τις, οικονομικέ ε, οικονομικές δραστηριότητες, ιδίως όσον αφορά τον παραδοσιακό ελευθερικό στόλο, όσον αφορά τους εργαζόμενους επίσης κατά τρίτο. Αυτό το οποίο θέλουμε είναι να στείλουμε ένα μήνυμα, ένα μήνυμα θετικό στο Μαρόκο και έτσι να πάμε σε ένα νέο πρωτόκολλο δίκαιο, ισορροπημένο και έτσι να έχουμε ανάπτυξη μιας βιώσιμης αλίας, αηφόρου που να ε, είναι συμβατό με όλων τα συμφέροντα. Ευχαριστούμε τον συνάδελφο Σάντζε Περσέντο. Ολοκληρώθηκε τώρα η διαδικασία Catch the Eye και θα δώσω το λόγο στην Επίτροπο κυρία Δαμανάκη. Ευχαριστώ. Πρέπει να δώσω κάποιε διευκρινήσει. Η Κομισιόν είναι εδώ για να υπερασπίσει τα κοινά ευρωπαϊκά συμφέροντα. Η κοινή αλληλευτική μας πολιτική υπερασπίζεται τα κοινά μας οικονομικά συμφέροντα. Δεν μπορώ να δεχθώ τα επιχειρήματα του τύπου ότι αυτή η συμφωνία είναι υπέρ ενός ή άντε δύο κρατών μελών που ψαρεύουν εκεί. Όλοι είμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση, όλοι καταναλώνουμε ψάρια. Είναι πολύ σημαντικό για τη διατροφή μας. Είμαστε οι πρώτοι καταναλωτές ψαριών στην, ε, στον κόσμο και θέλουμε καλές σχέσεις με όλους τους μεσογειακούς λαούς για να εξασφαλίσουμε αυτά τα ψάρια. Οι εποχές είναι χαλεπές, η, η κατάσταση είναι δύσκολη, αλλά δεν είναι σωστό να τα βλέπουμε τα πράγματα έτσι τόσο κοντόθωρα. Δεύτερη διευκρίνηση. Ναι, η Κομισιόν ενδιαφέρεται για τα δικαιώματα το, του λαού της περιοχής. Δεν είμαστε αδιάφοροι για τα, απέναντι στα δικαιώματα των, του, των Γι' αυτό ακριβώς έχουμε το διάμεσο πρωτόκολλο, γι' αυτό πιέσαμε την κυβέρνηση του Μαρόκου να μας δώσει στοιχεία για το κατά πόσον ε, και πώς θα υποφεληθεί ο πληθυσμός από την συμφωνία. Γι' αυτό έχουμε το διάμεσο πρωτόκολλο Γι' αυτό προσπαθούμε να διαπραγματευτούμε μια νέα συμφωνία και να λάβουμε υπόψη μας όλα όσα είπατε. Και αυτό που προσπαθούμε να πετύχουμε είναι ότι αν υπάρξει τελικά νέα συμφωνία που θα συμπεριλαμβάνει και τη Δυτική Σαχάρα, τότε θα υπάρχει μια προϋπόθεση ότι πραγματικά ο τοπικός πληθυσμός θα υποφεληθεί από αυτή τη συμφωνία όντως ενδιαφερόμαστε. Δεν είναι εύκολο να επιλύσουμε ένα διεθνές πρόβλημα μέσω μιας τέτοιας συμφωνίας. Και δεν μπορεί να δεχτεί μια τέτοια ιδέα η Κομισιόν. Ας είμαστε ξεκάθαροι λοιπόν. Είμαι εδώ, θα σας τα εξηγήσω όλα. Και θέλω να πω ότι η Κομισιόν θα σεβαστεί την ψήφο σας. Θέλω όμως να μου δώσετε μια ξεκάθαρη απάντηση. Θέλετε νέα συμφωνία σας υπόσχομαι ότι θα κάνω ό,τι μπορώ, ούτως ώστε η συμφωνία να είναι καλύτερη, αν υπάρξει. Καλύτερη συμφωνία σημαίνει ε, οικονομικά εποφελής, περιβαλλοντικά φιλική και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Σύμμορφη λοιπόν προς το διεθνές δίκαιο. Και αυτά όλα δεν είναι εύκολα. Δεν είναι τόσο εύκολα όσο φαίνονται. Δεν είναι εύκολο να σεβαστούμε το διεθνές δίκαιο στην προκειμένη περίπτωση. Αλλά θέλω να μου δώσετε μια ξεκάθαρη άποψη. Βλέπω ότι υπάρχουν διαφορετικέ απόψει μέσα στο Κοινοβούλιο. Υπάρχουν ορισμένοι που είναι εναντίον τη ίδια τη Αλλιευτική συμφωνία. Ορισμένοι ε, δεν θέλουν να υπάρξει καν συμφωνία. Ορισμένοι θέλουν συμφωνία, αλλά καλύτερη. Εντάξει, αλλά πέστε μα κι εσεί τι να κάνουμε τέλο πάντων. Θα ήθελα να τελειώνουμε τέλο πάντων. Μίλησα αρκετά. Εγώ σας είπα ότι η Κομισιόν ετοιμάζεται ήδη. Ετοιμάζει μια διαπραγματευτική εντολή για την επόμενη συμφωνία και σας βεβαιώ ότι η επόμενη συμφωνία θα είναι καλύτερη από τη σημερινή, αν θα την διαπραγματευτούμε τελικά, αλλά θέλουμε όμως γι' αυτό τη σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου. Γιατί αν το Κοινοβούλιο πει όχι στη συμφωνία, τότε δεν θα υπάρξει συμφωνία. Να το πούμε ξεκάθαρα. Και να μην προσπαθούμε να κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας. Θέλω να μου πείτε ξεκάθαρα τι να κάνω. Για το παρελθόν συμφωνώ μαζί σας. Οι παλιές συμφωνίες δεν ήταν οικονομικά επωφελείς, δεν ήταν οικονομικά περιβαλλοντικά φιλικές, γι' αυτό θέλουμε διαφορετική συμφωνία πια. Γι' αυτό θα υπάρξει μεταρρύθμιση. Και ελπίζω να μας υποστηρίξετε, ούτω ώστε να περάσει αυτή η μεταρρύθμιση από το Συμβούλιο. Αλλά γι' αυτό πρέπει να με βοηθήσετε και να με φωτίσετε. Εγώ πιστεύω ότι χρειαζόμαστε μια συμφωνία. Χρειαζόμαστε καλή συμφωνία, αλλά τη συμφωνία τη χρειαζόμαστε, γιατί αλλιώ ε, θα μείνουμε απομονωμένοι από, την από τον υπόλοιπο κόσμο. Ευχαριστούμε την Επίτροπο κύριε Δαμανάκη και δίνουμε το λόγο στον εισηγητή του κύριο Χάγκλουν για δύο λεπτά για να κλείσει αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε και όλοι μας είμαστε ικανοποιημένοι που θα προσπαθήσουμε να υπάρξει καλύτερη συμφωνία στο μέλλον. Αυτό δεν το αμφισβητούμε και αυτό θέλουμε. Δεν συμφωνώ με το συμπέρασμά μας όσο ότι πρέπει να υπερψηφίσουμε μια τρομακτική συμφωνία που σχεδόν όλοι θεωρούν ότι είναι κακή μόνο και μόνο για να, πετύχουμε την καλή ε, συμφωνία στο μέλλον. Δεν λειτουργεί έτσι το πράγμα. Η ευθύνη μα με βάση τη συνθήκη τη Λισαβόνα είναι να πάρουμε θέση για το τρέχον πρωτόκολλο. Δεν ψηφίζουμε για το επόμενο πρωτόκολλο. Γι' αυτό ψηφίζουμε για το τρέχον πρωτόκολλο, το οποίο είναι κάκιστο. Εγώ θα ψηφίσω υπέρ ένα τέτοιο ψυχικό πρωτόκολλο. Ε, Και σας πω, αγαπητοί φίλοι, αναφέρθηκε ότι αυτό το πρωτόκολλο πρόκειται να μας οδηγήσει σε δημιουργία θέσεων εργασίας. Όμως, 45.000 ευρώ κοστίζει σε επιδοτήσεις η κάθε τέτοια θέση. Είναι αυτό θέση εργασία, είναι αυτό σωστό για το προλογούμενο. Όχι, μόνο 15% έχει χρησιμοποιηθεί ε, ε, από τον, τον, τον... Ε, έχει ωφεληθεί το σώμα από του ψάδε στο Μάροκο αυτό, ούτε αυτό επομένω ισχύει ότι ωφελούνται αυτοί στο Μάροκο. Πάντω αυτή η διαρκή σχέση με το Μάροκο είναι πάρα πολύ σημαντική. Άρα υπάρχει τώρα μια τέτοια σχέση γνίαση ε, έτσι κι Είναι δεδομένη αυτή η πολιτική. Και όλα αυτά θα ισχύσουν διότι όλοι θέλουμε να υπάρχει μια τέτοια συμφωνία και επομένω ας προσοχή μα σε αυτή την κατεύθυνση αλλά πρώτα πρώτα να έχουμε ξεκάθαρη θέση ας είμαστε υπεύθυνοι στην ψηφορία μας όσον αφορά αυτή τη συμφωνία που δεν είναι η μέλουσα, είναι η σημερινή. Όσον αφορά τώρα τη Δυτική Σαχάρα, με μεγάλη μου χαρά διαπιστώνω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να βρει νέε ρυθμίσει, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι είναι πάρα πολλοί συνάδελφοι εδώ που θεωρούν ότι είναι προβληματική η ισχύουσα σημερινή ρύθμιση και πάρα πολλέ χώρε επίση. Αυστριακή, Σουηδή, τώρα η Bundestag, οι Ολλανδοί, οι Κύπροι έχουν επικρίνει. Γι' αυτό και υπήρχε πολύ σκληρή αναμετή στο Συμβούλιο. Δεν υπήρξε ομοφωνία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Χάγκλουντ. Ολοκληρώνεται λοιπόν η κοινή συζήτηση. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο στις 11.30 ε, και όχι την 5η. Επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η επομενο σημειο στην μεισια διαταξη ειναι η εκθεση του κυρίου Μπέργκε για την